η έκθεση του κυρίου Καπάτο με θέμα την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Το λόγο έχει ο εισηγητής κύριος Καπάτο ε, για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Σου... Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε την ευκαιρία τώρα να κάνουμε κάποιες προτάσεις Βέβαια, ο χρόνος πιέζει, αλλά επιτρέψτε μου να φέρω τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον, για το Συμβούλιο. Οι κυβερνήσει των κρατών μελών συνεδριάζουν με ε, νομοθετικές αρμοδιότητε. Και πάντα όταν κάποιο όργανο συνεδριάζει και έχει νομοθετικές αρμοδιότητες θα πρέπει να είναι δημόσιες η συνεδριάσεις του. Θα ήθελα να τονίσω το εξή εδώ και να υπογραμμίσω. Υπάρχουν βέβαια κάποιες τροπολογίες του ΕΛΚ που ζητούν ε, κατά τμήματα ψηφοφορίες για ορισμένα άρθρα. Ελπίζω να μην θέλουν να απαλείψουν σημαντικά σημεία της έκθεσης. Παράδειγμα, η παράγραφος 3, όπου η έκθεσή μου ζητά να δοθεί συνέχεια την υπόθεση Τούρκο, την απόφαση του ΔΕΚ που ήταν πρώην ευρωβουλευτής του ριζοσπαστικού κόμματος. Είχε δικαιωθεί ε, στο 10 ακριβώ ε, για ε, τον, να είναι δημόσια τα έγγραφα και γνωμοδοτήσει τη νομική υπηρεσίας των θεσμικών μας οργάνων. Το ίδιο ισχύει για την υποχρέωση Τη ταυτότητα τη αντιπροσωπεία των κρατών ε, μελών και τη τάση που τηρούν στο Συμβούλιο. Έχουμε το δικαίωμα να ξέρουμε ποια χώρα μέλο ψηφίζει τι στο Συμβούλιο. Ελπίζω να μην καταψηφιστεί και επαληφθεί η παράγραφος 3. Τα ίδια ισχύουν για την παράγραφο 9. Θα πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων, το λεγόμενο κορεπέρ. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τα έγγραφα τη συνεδρίαση να είναι δημόσια. Ας πούμε, τα έγγραφα που αφορούν τη διεθνή πολιτική δεν μπορεί να χαρακτηρίζονται ε, απόρριτα, διαβαθμισμένα τα έγγραφα αυτά. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό για το κοινοβούλιο μας. Εμείς θα πρέπει να είμαστε οι πρώτοι που θα έχουμε την πρόσβαση στα έγγραφα και θα δίνουμε πρόσβαση για το κοινό στα δικά μας έγγραφα με μητρώα, με τήρηση παρουσιών, απουσιών, ποιος βουλευτής είναι παρόν, ποιος είναι απόν, ποιος ψηφίζει τι. Επίσης και προφανώς ε, τι ε, οικονομικές απολαβές έχει ο κάθε βουλευτής θα πρέπει να αποφύγουμε το εξή σφάλμα. Γιατί και εδώ ζητείτε στην παράγραφο 5 ψηφοφορία κατά τμήματα. Μπορεί ορισμένες από τις πληροφορίε αυτές να είναι εμπιστευτικέ και να παραμένουν, και το λέω και προ την κυρία Σέλτσαρ αυτό, Εάν οι πληροφορίε αυτές, λέγω, ε, παραμένουν εμπιστευτικέ, παρέμεναν, τότε αυτό θα μας έκανε ακόμα περισσότερο ευάλωτους ε, δημαγωγικές επιθέσεις κατά των Ευρωβουλευτών. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εδώ συνάδελφοι που ε, έχουν μαγνητοσκοπήσει άλλους βουλευτές, που ε, κατασκοπεύουν ε, άλλους συναδέλφους. Το θέμα βέβαια δεν είναι απλώ να αποφύγουμε τέτοια φαινόμενα, αλλά να έχουμε πλήρη διαφάνεια στις εργασίες μα που να είναι δημόσιες και να μην έχουμε κάποιου που να μας ε, κατασκοπεύουν από την κλειδαρότρυπα. Α ανοίξουμε τι θύρε να μην υπάρχουν κλειδαρότρυπες και να βγάλουμε στο διαδίκτυο τι κοινοβουλευτικέ μα εργασίε και στην Ολομέλεια και στι επιτροπέ. Ένα τρίτο που θέλω να σα πω είναι πώ θα γίνει αυτή η πληροφόρηση. Στην παράγραφο 7 επίση ε, έχει ζητηθεί ψηφοφορία κάτι τμήματα από το ΕΛΚΑ ζητούμε να χρησιμοποιούνται έγγραφα ανοιχτής πηγής όπως λέγεται το κείμενο είναι ε, έτσι, ένας τεχνολογικός όρος με αποτελεσματική πολυγλωσία και τεχνολογίες που επιτρέπουν και σε άτομα με αναπηρίες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα όλα αυτά αναγράφονται στην παράγραφο υπεριθμών 7 ελπίζω να μην ε, διαφωνήσει κανείς για την πολυγλωσία ας πούμε στο κείμενο ανοιχτή πηγή. Ποιο μπορεί να διαφωνήσει για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες. Είναι θεμελιώδες αυτό για τους Ευρωπαίους πολίτες. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε, μάλλον η αρμόδια Επιτροπή ε, πρότεινα θεώρηση του κανονισμού μα τροποποίηση. Υπάρχει και έκθεση Κάσμα, θα τα ξαναπούμε αυτά. Αλλά η δική μου έκθεση είναι ένα πρώτο βήμα για να τεθεί το πλαίσιο αυτό και ελπίζω οι προσπάθειε αυτέ να μην αποβούν άκαρπε και να επιτύχουμε με την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λόγο έχει η κυρία Βάλστρομ. Thank you, Mr. President, ε, Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση αυτή που είναι καλά γραμμένη και ενδιαφέρουσα. Συγχαίρω τον εισηγητή. Πρόκειται για ένα θέμα σημαντικό κυρίως όταν μιλούμε για την αναθεώρηση του κανονισμού 1049 και λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που θα επιφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας αν επικυρωθεί αυτή η ε, πρόκειται για την αρχή του κανονισμού 1049 θα ήθελα να υπενθυμίσω ένα από τα θετικά στοιχεία της εφαρμογής του κανονισμού. Πώς δείχνουν τα ποσοτικά στοιχεία και όπως γνωρίζει το Κοινοβούλιο, τα θεσμικά όργανα έχουν δώσει μεγαλύτερη πρόσβηση σε εγγραφά Έχουμε δεσμευτεί να συνεχίσουμε να, να αυξάνουμε την ε, διαφάνεια. Μερικές συστάσεις βεβαίως της εισήγηση πηγαίνουν πολύ πιο πέρα από την εφαρμογή του κανονισμού 1049 και ε, μερικά από αυτά τα θέματα δεν συνδέονται με τις ε, δραστηριότητες της, ε, της Κομισιόν. Όλα αυτά σχετίζονται με το άνοιγμα προς τους πολίτες και αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό για την επικοινωνία και την διαφάνεια. Θα αναφερθώ σε μερικές από τις συστάσεις και τις αρχές διότι χρήζουν ε, εξέταση σχετικά με το θέμα, με την υπόθεση Τούρκο. Εμείς λαμβάνουμε υπόψη το θέμα αυτό για να αυξηθεί το άνοιγμα ε, σε σχέση με τα έγγραφα, αλλά βεβαίως ισχύει για την Κοσμισιόν και για όλα τα θεσμικά όργανα και η Κομισιόν βεβαιώνεται ότι κάθε αίτηση πρόσβασης να αξιολογείται ανάλογα με την περίσταση βάσει των παραμέτρων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το θέμα των κοινών ε, κανόνων και διαδικαστικών μέτρων ε, απαιτεί ιδιαίτερη ε, εξέταση, διότι μερικές διαδικασίες είναι μοναδικές για κάθε θεσμικό όργανο και αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ακόμα λίγο χρόνο η ε, σύσταση συγχώνευσης ε, του κανονισμού 1049 ε, και 354 για το άνοιγμα των ιστορικών αρχείων είναι κάτι το περίπλοκο για ιδιαίτερο λόγο, διότι το άρθρο 255 της Συνθήκης ΕΟΚ και το κανονισμός 1049 δεν ισχύουν για όλα τα θεσμικά όργανα και σώματα και αυτό θα πρέπει να αλλάξει αν τεθεί σε ισχύ η συνθήκη, διότι θα διευρυνθεί το δικαίωμα ε, πρόσβαση στα έγγραφα για όλα τα θεσμικά όργανα ε, και οντότητες. Σχετικά με ε, τις κρίσεις του Ombudsman, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη αυτή την παρατήρηση και όπως γνωρίζετε έχουμε ένα έγγραφο από τον Ιούνιο του 2002 και από τότε η Κομισιό έχει θεσπίθει ένα μητρό για τις διαδικασίες της επιτροπολογίας και για άλλες ομάδες και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξυγχρονίσουμε το συχνολογικό σύστημα που έχουμε. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη πάντοτε λαμβάνουμε υπόψη ε, την ε, αύξηση της κάλυψης από το μητρό να καλύπτει όσο δυνατόν περισσότερο το μητρό ε, θα πρέπει να γίνει αυτό και επίσης επιβεβαιώνουμε την δέσμευσή μας να αναπτύξουμε το δημόσιο μητρό ούτως ώστε να ενισχύσουμε την διαβάνεια. Ε, στο ψήφισμα αναφέρεστε στο θέμα της διαχείρισης ε, των εγγράφων και το σχέδιο Transjai. Υποστηρίζουμε την ιδέα ε, μιας τεχνολογικής πύλης για να, ε, για να διευκολύνουμε την πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα. Αυτό απαιτεί μια κοινή μεθοδολογία για να δούμε όλες τις πρακτικές ε, συνέπειες για την αναγνώριση και την παραπομπή σε έγγραφα. Και βεβαίως θα θέλαμε μια πύλη η οποία αναλαμβάνει λαμβάνει υπόψη όλα τα έγγραφα κάθε θεσμικού οργάνου. Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας για το θέμα αυτό. Για το σχέδιο TransGI επανέρχομαι στα όσα είπα στην απάντησή μου του Οκτωβρίου ότι θα είναι ανοιχτό το σύστημα αυτό το 2010 για το κοινό. Θα ήθελα να σχολιάσω για το θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Καταλαβαίνω τι, ε, τι επιδιώκεται, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων έχουμε ήδη μια μέθοδο εργασίας ε, για την ανταλλαγή μυστικών πληροφοριών, απορρίτων πληροφοριών και αυτό αναφέρεται ε, σε παράρτημα της Συμφωνίας Πλαισίου και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το θέμα ε, του να μοιράζονται πληροφορίες τα θεσμικά όργανα δεν έχει σχέση με την δημόσια πρόσβαση και είναι ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά η έκθεση αυτή και η συζήτηση είναι μια συμβολή χρήσιμη επίσης και για μια άλλη στιγμή όπου θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ευρύτερα το θέμα Είμαι ευγνώμων για τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου σχετικά με το ε, θέμα του ανοίγματο και της διαφάνειας ούτως ώστε να έχουν μεγάλη προτεραιότητα ε, σε προσεχές μέλλον όταν θα έχουμε μια, την επόμενη εβδομάδα μια ε, κοινή συνεδρίαση μεταξύ της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και του Κοινοβουλίου της Τσεχίας όπου θα είμαι και εγώ παρούσα θα εξεταστεί το θέμα και το θέμα της αναθεώρησης του κανονισμού 1049. Δεν πρέπει η συζήτηση να λήξει εκεί. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε προόβουλα για ε, την νομοθεσία και για την διαφάνεια για τα μητρώα, να τα να είναι πιο φιλικά ε, για μια ενεργό διανομή και για μια ε, ταχεία δημοσίευση εγγράφων κάτι που έκανα πέρσι, έκανα το μητρό για την δική μου αλληλογραφία προσβάσιμο ε, στο διαδίκτυο και ελπίζω όλοι να έχετε παρόμοιες ιδέες για το τι μπορεί να γίνει ε, για να προωθήσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βάλστρο. Ακολουθούν οι ομιλητές εξ των πολιτικών ομάδων. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για δύο λεπτά το λόγο ο κύριος ε, Λοή Σερέρο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Καπάτο, η έκθεσή σας είναι γεμάτο καλές προθέσεις και είναι προφανέστατο ότι δεν χρειάστηκε καμία τροπολογία από ό,τι φάρηκε στην Επιτροπή Ελευθεριών. Εσείς ο ίδιος κάνατε 18 ολόκληρες τροπολογίες στην ίδια σας την έκθεση. Και τελικά Αυτές οι τροπολογίες έκαναν πιο ακραία την έκθεση. Αυτό εμένα με κάνει να αμφιβάλλω πάρα πολύ σοβαρά. Θα ήθελα να τις χωρίσω σε τέσσερις κατηγορίες, τις τροπολογίες που βάλατε εσείς ο ίδιος, στη δική σας έκθεση, την οποία στην αρχή όλοι υποστήριξαν είναι ανέφικτα τα πράγματα που ζητάτε. Κύριε Καπάτο, για παράδειγμα, ζητάτε πράγματα που δεν έχουν νομική βάση. Α πούμε, αν δεν τεθεί σε ισχύ ακόμα η συνθήκη τη Λισαβόνα δεν μπορούμε να εναρμονίσουμε κανονισμού διαφόρων επιτροπών. Αυτό που είπε και η Επίτροπος μόλις. για παράδειγμα, ζητάτε το έτο 2009 να διακηρυχθεί έτος της διαφάνειας. Μα είμαστε καταϊδρωμένοι και τελευταίοι, πολύ αργά. Ε, Με τα διάφορα πράγματα προς αποφυγή. Ζητάτε διαφάνεια στη συνεδριάση των πολιτικών ομάδων. Γιατί η ιδιωτική ε, στάση και ζωή είναι δικαίωμα. Αυτό δεν είναι έλλειμμα διαφάνειας. Αν εγώ θέλω να ε, απομακρυνθώ από το πολιτικό μου κόμμα ή την πολιτική μου ομάδα, στις πολιτικές ομάδες θα πρέπει να είναι ε, προστατευμένες ιδιωτικές συζητήσεις. Δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω. Κάποια άλλα που ζητάτε είναι γκρίζες ζώνες. Λέτε ότι το 90% το νομοθετικών ε, ε, δραστηριοτήτων είναι επιτροπολογία. Μα υπερβάλλεται. Τι θέλουμε εμείς και άλλους μηχανισμούς και άλλη γραφειοκρατία και άλλους ελέγχους. Εις βάρος της διαφάνειας είναι αυτό που θέλουμε τελικά να έχουμε. Και η διαφάνεια σημαίνει απλές διαδικασίες. Και τέλος, πριν αρχίσει να μου φωνάζει ο πρόεδρος, υπάρχουν και διάφορα πράγματα άχρηστα, περιτά. Για παράδειγμα, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ ελκυστικό και τη μόδα για την κοινή γνώμη να λέμε δραστηριότητε των βουλευτών με διαφάνεια. Ξέρουμε ποιοι παρευρίσκονται στη Ολομέλεια. Μα τα ξέρουμε αυτά, κύριε ε, Καπάτο. Και στι επιτροπέ υπογράφουμε, τα ξέρουν και οι πολίτε. Και τι λεφτά παίρνουμε, τα ξέρουν τα, τα, την ημερήσια αποζημίωση και γενικά τι απολαυέ μα. Υπάρχει πρόσβαση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ ε, τη μόδα και μα τιμά και μα ε, κοσμεί το να ασχολούμαστε με τη διαφάνεια, αλλά να βλέπουμε τα πράγματα όπως έχουν. Αυτό είναι η διαφάνεια. Και όταν τα δείχνουμε από άλλο πρίσμα, κύριε Καπάτο, αυτά δεν είναι διαφάνεια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σα. Τίποτα. Καλωσύνη σα. Λοιπόν, πάμε στου σοσιαλιστέ τώρα για δύο λεπτά. Ο κύριο Κάσμαν. Uh, σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Μάρκο, για την εξαιρετική έκθεση. Δυστυχώς θα συμφωνήσω με ορισμένους άλλους ότι κάπως ξέφυγες λίγο από το θέμα. Και ξέρω και γιατί. Ο προηγούμενος ομιλητής είπε ότι είναι αδύνατον, αδύνατο να γίνουν αυτά τα πράγματα. Μα ακριβώς αυτό. Πρέπει να ζητούμε τα αδύνατα ώστε να πετύχουμε κάποια πράγματα. Ε, οι ευρωβουλευτές να βάζουν στους ιστοσελίδες τους πληροφορίες για το τι κάνουν και πού πηγαίνουν δεν σημαίνει ότι αυτά τα πράγματα είναι και αποτελεσματικά και καλά. Ο οργανισμός έχει σχέση με την πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα τα οποία διαθέτουν ή παράγουν τα τρία θεσμικά όργανα όταν λειτουργούν υπό την νομοθετική τους λειτουργία. Αυτό, σε αυτό πρέπει να επανέλθουμε. Πρέπει να εξετάσουμε και να ορίσουμε τι είναι νομοθετική λειτουργία. Και πρέπει να βελτιώσουμε το όσο έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα. Εγώ αυτό επιθυμώ να κάνω σε συνδυασμό με τις προσπάθειες όλων των υπολείπων και Καλωσορίζω την ε, Σουηδή Υπουργό, κυρία Σίλια Μάλστρομ, η οποία έχει κάνει σχετική προσπάθεια και θέλουμε να προωθήσουμε ολόκληρη αυτή την υπόθεση της πρόσβασης. Γιατί? Διότι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν ότι συμβαίνουν πράγματα, ιδίω στο Συμβούλιο Υπουργών όπου ε, βλέπουν οι πολίτε του εθνικού του υπουργού να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Υπουργών και να λαμβάνουν αποφάσει, αλλά δεν γνωρίζουν τι συζητούν και πώ συζητούν. Θέλουμε λοιπόν εμείς να δείξουμε πώς ψηφίζουν οι ε, ε, ε, υπουργοί και αυτοί τότε θα είναι υπόλογοι στους ψηφοφόρους τους στις χώρες μέλη και τότε πια οι πολίτες θα θεωρήσουν ότι ναι έχουμε κάποια σχέση με τα όσα συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς λοιπόν υπερεύεις τα όρια αγαπητέ Μάρκο. Αν δεν έλεγες από την αρχή ότι είσαι Ιταλός ριζοσπαστικός δεν θα το πίστευα ποτέ αλλά δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τα πολιτικά κόμματα να ε, ανοίξουν τις ε, εσωτερικές τους συζητήσεις. Δεν πρόκειται ποτέ να το δεχθούν αυτό το πράγμα, όπως το εξήγησε και ο προηγούμενος ομιλητής. Εμείς πιστεύουμε σε μια Ευρώπη που είναι υπόλογη στους πολίτες της. Η ε, λίστα ψηφοφοριών λοιπόν θα είναι δύσκολο να γίνει για τις τροπολογίες σου, πράγματι. Η καρδιά μου είναι μαζί σου, αλλά πρέπει να ακούσω το μυαλό μου. Ευχαριστώ για δύο μισή λεπτά από του φιλελευθέρου, ο κύριο Άλβαρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλώ όρισατε. Αύριο θα ψηφίσουμε την έκθεση του συναδέλφου Μάρκο Καπάκτο για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα και ο Μάικλ Κάσμα που είναι καλό συνάδελφο και εξαιρετικά αποτελεσματικό είπε ότι θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο κοινό ε, στα έγγραφα που συζητούνται εδώ και αποφασίζονται. Όπως είπε ο κύριος Ερέρο ή ο ε, Κλικάσμα, μπορούμε να προσάψουμε στο Μάρκο ότι υπερβάλλει, αλλά δεν νομίζω να ευσταθεί αυτό. Η συζήτηση για το αν ε, καταρχήν θα πρέπει να είναι δημόσια η συνεδρία των πολιτικών ομάδων μπορεί να συζητηθεί. Δηλαδή αν το επιθυμούν ορισμένα ε, μέλη, η πλειοψηφία των μελών μπορεί να είναι και κλεισμένο το θύρο Το ξέρουμε όλοι. Στι συνεδριάσει μα υπάρχουν θέματα που πρέπει να λύσουμε στο εσωτερικό τη πολιτική ομάδα και στο κάτω-κάτω ε, τα άπλητά μα δεν τα βγάζουμε στη φόρα. Το ίδιο ισχύει και για τα πολιτικά κόμματα, όχι πολιτικές ομάδες. Πάντα έχουν συμφέρον να υπάρχει κάποια διαφάνεια όταν τους εξυπηρετεί κομματικά. Αλλιώς δεν θα είχαμε ποτέ συνέδρια των κομμάτων που να τα δίδονται τόσο πολύ στη τηλεόραση και γενικά και ενδιαφέρον είναι αυτό. Κανένας δεν διαμαρτύρεται ε, και σε περιπτώσεις που μπορεί τα πνεύματα να θερμαίνονται. Μπορώ να πω λοιπόν γενικά ότι ο Μάρκο έχει κάνει καλή δουλειά εδώ Ακόμα και αν έχονται προτάσεις για βελτίωση από άλλες πολιτικές ομάδες που το έχουμε συνηθίσει. Καμιά φορά είναι και τόσο καλές που καλό θα ήταν να τις συζητήσουμε και να σκεφτούμε. Σε σύγκριση όμως με τα άλλα δύο θεσμικά όργανα, το Κοινοβούλιο μπορεί να θεωρηθεί πρωτοπόρο, όπως και στο παρελθόν, για τη διαφάνεια. Και... Ε, ακριβώς για την πρόσβαση στα έγγραφα και τη διαφάνεια των συνεδριάσεων και των δραστηριοτήτων των Ευρωβουλευτών είμαστε πολύ πιο ανοιχτοί από οποιαδήποτε άλλη Εθνική Βουλή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν επιδεχόμαστε βελτιώσει σε άλλα θεσμικά όργανα, ιδιαίτερα στο Συμβούλιο, που δυστυχώ αυτή τη στιγμή απουσιάζει. Το είπε και ο Μάικλ προηγουμένω. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο πήρε ποια απόφαση και με ποιο τρόπο στο Συμβούλιο για να ε, έχουμε και υπεύθυνη πολιτική δράση και στάση. Ακόμα πιο σημαντικό είναι η πρόσβαση στα έγγραφα να είναι δεδομένη. Για παράδειγμα, στα πλαίσια τη διαδικασία επιτροπολογία. Ιδιαίτερο παράδειγμα ήταν ο κανονισμός για ε, τα υγρά ε, στις χειραποσκευές, όπου το παράρτημα δεν ήταν ε, δημόσιο, δεν μπορούσε να το κοιτάξει κανείς ούτε ευρωβουλευτής. Και τελικά επιβλήθηκε να μπορεί το κοινό να έχει πρόσβαση, να καταλαβαίνει, να ξέρει τι γίνεται και ενδεχομένω να αλλάζει και τακτική σε εκλογέ. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μου δώσατε. Καλή τύχη Μάρκο αύριο στην ψηφοφορία και νομίζω ότι θα το φέρουμε σε αίσιο πέρα. Σε ευχαριστώ. Την ε, Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Τσενέσκι. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίε και κύριοι. πρέπει να μας απασχολεί περι, περισσότερο αυτοί που βρίσκονται εκτός, οι άνθρωποι εκτός και όχι να έχουμε μια Ευρώπη από και για τους ευρωκράτες και για το σκοπό αυτό πρέπει να αυξήσουμε τη διαφάνεια και επίσης την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων. Νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι δεν ρωτούμε τους άλλους ποιες είναι οι απόψεις τους. Ε, και δεν, ε, δεν χρησιμοποιούμε και τις δημοψηφίσματα για να δούμε ε, τι σκέφτονται οι άλλοι. Ίσως αυτό είναι έχει σχέση με το θέμα ότι δεν δημοσιοποιούμε τις εργασίες των επιτροπών, των ομάδων. Πρέπει να έχουμε αυτόματη ανοιχτή πρόσβαση στις πληροφορίες τους, ώστε οι εκτός να ξέρουν πού να απευθυνθούν για να βρουν τις πληροφορίες που θέλουν. Υπάρχει ένα επιχείρημα ότι το, βρίσκονται τα θεσμικά όργανα πολύ μακριά από τους πολίτες. Πρέπει να κάνουμε κάτι για να αντιστρέψουμε αυτή την άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Από την Ενωτική Αριστερά και τη Βόρεια Αριστερά για ένα λεπτό. Η κυρία Σουένσον. Ευχαριστώ ε, και ο κύριος Καπάτο δείχνει στην έκθεσή του ότι υπάρχουν πολλά κενά, πολλές ελλείψεις σχετικά με το δημόσιο χαρακτήρα και της διαφάνειας. Είμαι υπέρ μιας μεγαλύτερης διαφάνειας και υπέρ των τροπολογιών που παρουσίασε ο ίδιος ο εισηγητής. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να είναι πράγματι υπέρ μιας μεγαλύτερης διαφάνειας και νομίζω ότι η έκθεση του κυρίου Κασμάν επίσης θα υιοθετηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι απαράδεκτο να εξουσιοδοτούμε κατά κάποιο τρόπο ε, την ομοθεσία, διότι κάθε χρόνο Υιοθετούμε μερικές πράξεις ε, νομοθετικές που δεν είναι αυτόματα διαφανείς. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια σχετικά με την συμμετοχή των Ευρωβουλευτών σε εργασίες της Ευρωκοινοβουλίου και ε, σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντα στο Ευρωκοινοβούλιο των διαφόρων Ευρωβουλευτών. Όλα αυτά υπέρ της διαφάνειας. Είμαι υπέρ επίσης των δημοσίων μητρώων. Δεν πρόκειται εδώ για μια απέτηση λαϊκίστικη, πρόκειται για μια απέτηση πολιτική. Ο κύριος Λούγκρεν, δύο λεπτά. Κύριε ε, Πρόεδρε, είναι σημαντικό για κάθε δημοκρατία αυτό. Στη δημοκρατία οι ψηφοφόροι διαλέγουν, εκλέγουν αυτούς που θα τους εκπροσωπούν και θα λαμβάνουν αποφάσεις στο όνομά τους. Είναι παράλογο αυτοί οι εκλεγμένοι εκπροσωποί τους να μην δίνουν πληροφορίες σε αυτούς που τους εξέλεξαν. Αυτό όμως γίνεται συχνά και για πολλούς λόγους κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, πολύ συχνά ε, αναθέτουμε την εργασία σε άτομα που δεν έχουν εκλεγεί και μετά επιθυμούμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια λένε, αλλά για να γίνει αυτό υπάρχουν εξαιρέσεις, παρεκκλήσεις από αυτή τη διαφάνεια. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να επανέλθουμε σε όλες αυτές τις ιδέες, τις έννοιες. Σήμερα δεν μπορούμε να κρατάμε μυστικές, απόρριτες ορισμένες πληροφορίες. Επιπλέον, οι πολίτες έχουν απαιτήσεις νόμιμες και δεν μπορούμε πλέον σήμερα να κρυβόμαστε πίσω από ορισμένε αφορμές ε, για να κρατούμε μυστικές πληροφορίες. Παλιότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πάντα ήταν απόρριτα. Ακόμα και το όνομα ε, των επιτρόπων, αλλά σιγά σιγά άρχισε να ανοίγεται προς τα έξω η Ένωση. Ορισμένα σημαντικά βήματα έγιναν από το 1993 και μετά το 1998 έγινε δεκτή μια μεγαλύτερη διαφάνεια και με κάποια υπερηφάνεια διαπιστώνω ότι η χώρα μου, η Σουηδία είναι αυτή που έχει την μεγαλύτερη παράδοση διαφάνειας των δημοσίων εγγράφων. Είναι σημαντικό επίσης η υπόθεση Τούρκο ε, να την παρακολουθήσουμε μετά την απόφαση που λήφθηκε πέρσι το καλοκαίρι αλλά έχει απομείνει ακόμη πολλής δρόμος αν θέλουμε η διαφάνεια να επικρατήσει πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλά εμπόδια ακόμα, γι' αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε την εισήγηση του κυρίου Καπάτο που είναι μια αρχή σε αυτόν τον μακρύ ε, δρόμο. Ρωμανιολό, ένα λεπτό. Είναι λίγα δευτερόλεπτα για να πω ότι συμμερίζομαι ένα μεγάλο μέρος ε, των συμπερασμάτων του συναδέλφου Καπάτο δεν μπορεί να γίνει αλλιώ, διότι νομίζω ότι είμαι ο μόνος Ιταλός Ευρωβουλευτής που προσπάθησε ε, να δημοσιεύει κάθε ε, χρόνο στο Μητρό της δραστηριότητες μου, τις κοινοβουλευτικές και τον κατάλογο των θεμάτων, των ερωτήσεων και απαντήσεων από τους Ιταλούς Ευρωβουλευτές εδώ θα ήμουν περισσότερο ευχαριστημένος αν ο Ιταλικός ε, τύπος θα είχε απηχήσει αυτά. Ίσως τον Ιταλικό τύπο μπορούμε να τον κατακρίνουμε για άλλα πράγματα, αλλά αν μπορούσε να μεταδίδει τις δραστηριότητες των, Ευρωπαίων, ε, των Ιταλών Ευρωβουλευτών εδώ θα ήταν αυτό χρήσιμο και θα μπορούσε να δείξει μέχρι ποιου βαθμού οι δραστηριότητες οι κοινοβουλευτικές αν διεκπεραιώνονται καλά είναι ανεξάρτητες από τις άλλες νομοθετικές αρχές. Επικροτώ λοιπόν την πρωτοβουλία του Μάρκο ε, και θα ψηφίσω περίπου όλα τα σημεία της ε, εισήγησής του. Ευχαριστώ Μενέσκου, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αρχή της διαφάνειας. Γίνεται αναφορά στο πρώτο και έκτο άρθρο της συνθήκης και στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέλησε πάντοτε με τον πλέον διαφανή τρόπο να λαμβάνει αποφάσεις ώστε να είναι πιο κοντά στους πολίτες. Το Κοινοβούλιο δεν είναι το μόνο που θέλει το κοινό να έχει ε, πρόσβαση στα έγγραφα διότι αυτό αυξάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι καλή η πρόσβαση για την ώρα, αλλά είναι προφανές ότι η νομοθεσία ευρωπαϊκή του 2001 για την ρύθμιση αυτής της πρόσβασης πρέπει να ε, επικαιροποιηθεί. Γι' αυτό ζητήσαμε προτάσεις ε, για την αναδιατύπωση ε, του εγγράφου αυτή, ούτως ώστε όλα τα έγγραφα να είναι διαθέσιμα για το κοινό. Η Κομισιόν έλαβε υπόψη τις συστάσεις αυτές που περιλήφθηκαν στη νέα πρόταση κανονισμού του 2008. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων υπήρξαν διστάμενες απόψεις και ε, οι διαπραγματεύσεις οδήγησαν στην καλύτερη δυνατή απόφαση για όλους. Ο πολίτης πρέπει να ενημερώνονται κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαδρομής, ε, διότι οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα τη ζωή τους. Ευχαριστώ. Νίκο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η διαφάνεια και η δημοσιότητα έχουν ιδιαίτερο βάρος τώρα όπου πλησιάζουμε στις ευρωεκλογές. Πρέπει να διασφαλίσουμε την μέγιστη δυνατή συμμετοχή του κοινού στις εκλογές. Εάν μπορέσουμε να παρουσιάσουμε πληροφορίες σε κατανοητή γλώσσα στους πολίτες, θα τους προκαλέσουμε και το ενδιαφέρον και των μεγάλων και των μικρών και των πλέον ηλικιωμένων δηλαδή. Θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους κριτήρια μέσω των οποίων να μπορούν να αναζητήσουν στο διαδίκτυο ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος των ευρωβουλευτών που ψηφίζουν, πώς ψηφίζουν, πώς εργάζονται στις επιτροπές ή τις αντιπροσωπείες. Να έχουν μια πλήρη εικόνα δηλαδή του έργου μας. Εγώ είμαι επίσης υπέρ της ιδέας της ε, δημιουργίας ενός κοινού διαθεσμικού αρχείου ε, των εγγράφων που να υπάρχει και εκεί πρόσβαση και να είναι ένα one-stop shop για όλα τα έγγραφα. Εν τέλει υποστηρίζω την έκθεση του κ. Καπάτο. Η κυρία Χάρκιμ Συγχαίρω τον Μάρκο Καπάτο για την έκθεσή του και πολύ καλά κάνουμε που τη συζητούμε τώρα εδώ. Όταν μιλούμε για ε, το να είναι υπόλογοι βουλευτές για διαφάνεια κλπ. Είναι πολύ σημαντικό και για μας. Έχω ορισμένες επιφυλάξεις βέβαια. Εάν θέλουμε να δώσουμε πληροφορίες για τις δραστηριότητες των ευρωβουλευτών, πρέπει οι πληροφορίες αυτές να είναι κατανοητές διότι αλλιώς το υποβαθμίζουμε. Είναι πολύ ευρύ αυτό. Δεν είναι μόνο το θέμα της παρουσίας των βουλευτών στις επιτροπές και στην Ολομέλεια. Και αν δώσουμε πληροφορίε για τους βουλευτές και το έργο τους, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πτυχές του έργου, του, του έργου τους. Και έρχομαι στα όσα είπε ο κύριος Ρωμανιόλη, που είπε ότι η καλή δουλειά που γίνεται εδώ δεν ε, βρίσκει απήχηση στα μέσα μαζική ενημέρωση. Μα τα μέσα μαζική ενημέρωση ενδιαφέρονται μόνο όταν κάποιο δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Συμφωνώ με τον Μάικλ Κάσμαν ότι όλοι οι πολίτε θα πρέπει να γνωρίζουν με ποιο τρόπο ψηφίζουν οι υπουργοί του στο Συμβούλιο Υπουργών. Διότι αλλιώ βεβαίω ρίχνουμε νερό στον μήλο εκείνων που μέμφονται τι Βρυξέλλε για οτιδήποτε άσχημο συμβαίνει στι πατρίδε του. Ο κύριο Μάρτιν ένα λεπτό. Η εμπειρία μου είναι πιθανώς πολύ παρόμοια με εκείνες εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Ήρθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1999 με, μεγάλη, με μεγάλο ενθουσιασμό που δεν δικαιολογήθηκε μετά. Έκανα λοιπόν κάτι που ήθελα, θέλω να κάνουν πολλοί πολίτες. Θα ήθελα να μάθω. Δηλαδή πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, πού πάνε τα λεφτά. Η ψηφοφόροι μου μου είπαν ότι δεν ξέρουμε τι κάνει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ δεν ήξερα. Και καταλήγω δυστυχώς στο, στην εμπειρία ότι πίσω από πολλά μέτρα κρύπτεται η πρόθεση να καλυφθούν, να συγκαλυφθούν ορισμένα πράγματα, να μην φαίνεται καθαρά ποιος είναι υπεύθυνο γιατί. Εγώ σας ενθαρρύνω να προχωρήσετε πολύ περισσότερο και από εκεί που προχωρεί η έκθεση καπάτων και να δοθεί αυτή η πληροφορία σε όλους τους τομείς, σε όλα τα επίπεδα. Και τα λέω αυτά μετά από 10 χρόνια εμπειριών εδώ. Κοέλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αρχή της διαφάνειας είναι θεμελιώδης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενισχύει τον δημοκρατικό χαρακτήρα των θεσμικών μας οργάνων, επιτρέπει την συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και εξασφαλίζει μεγαλύτερη νομιμοποίηση των θεσμικών οργάνων αφού αυτά είναι υπόλογα απέναντι στους πολίτες. Κάθε θεσμικό όργανο έχει και το καθήκον να ανοίγει τα έγγραφά του. Η δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα είναι βασικό θέμα για την αξιόπιστη ε, διασύνδεση και άλληλο συνεργασία των ε, θεσμικών οργάνων. Το Συμβούλιο έχει διακόψει την πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα και προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και η απόφαση στην ε, ε, υπόθεση Τούρκο. Υπάρχει και γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου Υπουργών που ζητεί το άνοιγμα, προτείνει τέλο πάντων το άνοιγμα ορισμένων εγγράφων σε διοικητικές διαδικασίες εξακολουθούν και υπάρχουν αδυνατά σημεία τα οποία πρέπει να αποκαλυφθούν και πρέπει να ενσωματωθεί η ε, απόφαση του ΔΕΚ για την υπόθεση Τούρκο. Ορισμένες προτάσεις του εισηγητού υπερβαίνουν τα όρια της νομικής βάσης. Τα είπαν αυτά οι κύριοι Ερέρο και Κάσμαν. Υπάρχουν διατάξεις για παράδειγμα που αναφέρονται χωρίς να υπάρχει καμία νομική βάση. Στην υπόθεση Τούρκο το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναγνωρίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί μια ισορροπία ανάμεσα στους κινδύνους που ε, συνεπάγεται η ε, δημοσιότητα ενός εγγράφου και στην ανάγκη να προστατευτεί η ε, πρόσβαση των πολιτών. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής γεγονός. Ο κύριος Καπάτο στην αρχή υποστηρίχθηκε από πολλούς συναδέλφους. Στη συνέχεια όμως έκανε ο ίδιος 18 τροπολογίες στην έκθεσή του, οι οποίες δεν γνώρισαν την υποστήριξη των συναδέλφων. Χρειάζεται όμως περισσότερη διαφάνεια στις εργασίες μας για να έχουμε και εμπιστοσύνη στα μάτια των πολιτών. Η ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημοσιεύει τα στοιχεία με τις δραστηριότητες του κάθε βουλευτού. Θα μπορούσε, ας πούμε, εκεί να συμπεριλαμβάνεται και ε, το είδος και ο αριθμός των τροπολογιών που έχει καταθέσει ο βουλευτής στην εγκάστοτε έκθεση για να βλέπουν οι πολίτες πώς συμβάλλουν οι βουλευτές ε, στη λήψη των αποφάσεων κτλ. Επίσης, άλλα θεσμικά όργανα θα πρέπει να δημοσιοποιούν τις δικές τους ε, συνεδριάσεις, το Συμβούλιο, πριν τεθεί σε ισχύ υποχρεωτικά από τη συνθήκη της Αφώνας. Το μας έσκαγε ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, οι πολίτες μεταξύ άλλων δικαιωμάτων έχουν και το δικαίωμα να γνωρίζουν τι κάνουν οι αιρετοί τους εκπρόσωποι και πώς ε, ασκούν τα καθήκοντά τους συγκεκριμένα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Συμβούλιο. Διότι τα έγγραφα του Συμβούλου είναι πάρα πολύ δύσκολα να τα βρει κανείς τα προγράμματα ενημερωτικά ε, στο διαδίκτυο θα πρέπει να είναι καλύτερα και πιο φιλικά προς το χρήστη, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να φτάνουν πιο γρήγορα στα έγγραφα. Αφήστε δε που δεν έχουν όλη τη δυνατότητα προσφυγή στο διαδίκτυο, όσο και αν είναι δεδομένο αυτό το μέσον σήμερα. Θα πρέπει να υπάρχουν και δημοσιεύσεις ε, γραπτές σε βιβλιοθήκες και να μπορεί κανείς να παραγγέλει διάφορα έγγραφα, διάφορα κείμενα και για ανθρώπους με αναπηρίες που δεν μπορούν ε, έτσι εύκολα να μπουν στο διαδίκτυο. Το θέμα των πολιτικών ομάδων όμως δεν είναι βέβαια θα πρέπει να δημοσιεύεται. Κυρία Σέντερσολτ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η διαφάνεια είναι ευρύ πεδίο και θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γνώρισε μεγάλη εξέλιξη. Νομίζω δεν θα διαφορήσει κανείς. Από τη θέση σε ισχύ ας πούμε του κανονισμού 1049 ε, και τις ιστοσελίδες στο διαδίκτυο έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες. Τα τελευταία χρόνια επίσης είδαμε δράσεις πολύ ενδιαφέρουσες από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα πράγματα δεν ήταν πάντα εύκολα, αλλά η συνεργασία μας νομίζω τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά καλή. Είναι πολύ καλή. Και θα πρέπει να το λέμε και αυτό όταν κάνει κάτι καλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τις το αναγνωρίζουμε. Βεβαίως είναι γεγονός, τα είπε και ο κύριος Άλβαρο προηγουμένως, ότι τίθεται το θέμα των ε, νομοθετικών ε, αποφάσεων και των ε, συζητήσεων που δεν είναι πάντα δημόσιες. Και έχει σημασία να γνωρίζουμε τι γίνεται στο Συμβούλιο, ας πούμε. Δεν λέω καθημερινά να έχουμε πλήρη αναφορά στα πρακτικά, ούτε χρειάζεται κάτι τέτοιο. Αλλά να έχουμε μια γενική εικόνα και μια γενική πληροφόρηση. Γενικά είμαι υπέρ τη πρόταση Καπάτο χωρίς να σημαίνει αυτό επιβάρηση. Ο κύριος Ρογκάλσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι τα δημοκρατικά συστήματα που βασίζονται σε ένα κράτος δικαίου σημαίνουν ότι τα όσα αποφασίζονται για τους πολίτες θα πρέπει να είναι δημόσια και να είναι υποχρεωμένα τα θεσμικά όργανα να το πράττουν αυτό ε, για τη διαφάνεια. Δηλαδή, να είναι δημόσιες οι συνεδριάσεις και οι ψηφοφορίες και τα σχέδια νόμου ακόμα. Δυστυχώς το Συμβούλιο δυσκολεύει την πρόσφαση σε ε, έγγραφα και αυτό εμποδίζει τους πολίτες να λαμβάνουν γνώση των κειμένων αυτών. Είναι πολύ σημαντικό όμως να ξέρουν οι πολίτες τι γίνεται, ειδικά στο διαδίκτυο. Χρειάζεται ε, μια ενιαία δικτυακή πύλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για τα έγγραφα, για τις διαδικασίες και για τα θεσμικά όργανα. Να έχουμε κοινού κανόνες για τις διοικητικές διαδικασίες, για την τήρηση κάποιων απορρίτων, τη διαβάθμιση των εγγράφων. Και παράδειγμα είναι το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντόιλ. Uh, Ευχαριστώ. Άκουσα προσεκτικά τον εισηγητή. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Πρόσβαση στο νομοθετικό έργο και πρόσβαση στα έγγραφα μη νομοθετικού έργου. Για το πρώτο, συμφωνώ αυτή την ενεργό διαφάνεια να είναι ο κανόνας. Να μειωθούν πολύ τα μη ανοιχτέ συζητήσει και συνεδριάσει του Συμβουλίου, ώστε να μπορούν να είναι υπόλογοι οι Υπουργοί. Και να σταματήσει επιτέλου αυτό που ακούγεται και σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια, που όλοι μέμφονται τι Βρυξέλλες, ενώ οι δικοί του Υπουργοί έχουν λάβει τι αποφάσει. αφού άλλωστε αυτοί εκλέγονται από του πολίτε. Από την άλλη μεριά να πούμε ότι όλε οι κοινοβουλευτικέ ομάδε ή όλε οι κομματικέ συνεδριάσει πρέπει να είναι ανοιχτές ε, ε, ε, στο κοινό, αυτά είναι ανοησίε. Εγώ δεν φοβούμαι τη διαφάνεια. Εμεί είμαστε έντιμοι άνθρωποι εδώ και μπορούμε να αρθώσουμε το παράστημά μα όταν πρόκειται για την αξιοπρέπεια του επαγγελματό μα. Ευχαριστώ. Κύριε Φατούτσο, εσεί τώρα. Sono assolutamente certo che... Ε? Ναι, ο συνάδελφός μας Καπάτο εκπώνησε μια εισήγηση και είμαι βέβαιος ότι έχει αποφύγει να καταπατήσει τα δικαιώματα των υπαλλήλων οι οποίοι ε, προσπαθούν να επιτελέσουν το καθήκον τους και να διαφυλάξουν το απόρριτο για ορισμένες ε, καταστάσεις ε, που οφείλουν να παραμείνουν απόρριτες από τη φύση τους. Αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό για να εγκριθεί αυτή η εισήγηση, αλλά θα ήθελα να αντιστρέψω τις ανησυχίες ορισμένων από εμά που έχουν εκφράσει ορισμένους φόβους. Φοβούνται ότι ε, το ε, δικαίωμα επιφύλαξης και το απόρριτο θα θυγούν. Τι συμβαίνει όταν ένας υπάλληλος ε, θέλει να μάθει τι κάνουμε εμείς οι άλλοι πολίτες. Δεν υπάρχει ε, μυστικό ε, σε ορισμένα κράτη, υπάρχουν, ακούνε ε, ακόμα τις συνδιαλέξεις, τις τηλεφωνικές, γίνονται υποκλοπές, τις συνδιαλλαγές ανάμεσα στη γυναίκα και τον άντρα της, τον πατέρα και το παιδί του. Ορισμένοι θέλουν να μάθουν γιατί υιοθετούνται ορισμένοι νόμοι, κανόνες και αποφάσεις νομοθετικές του κοινοβουλίου μας. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Ναι, το θέμα της διαφάνειας του ανοίγματος είναι θέμα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολούν σε σχέση με τόσα γίνονται στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτών των θεσμικών οργάνων. Θα, θα είναι ευκολότερο για αυτούς που βρίσκονται έξω και για τους ε, πολίτες, τους απλούς πολίτες να καταλάβουν τα όσα γίνονται εδώ. Νομίζω ότι υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης και μου φαίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε ε, να ε, τα διορθώσουμε τα πράγματα, να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Τα θεσμικά όργανα έχουν μια κρίση εμπιστοσύνης ε, και αυτό είναι το νόημα των δημοψηφισμάτων που είδαμε στην Γαλλία, στις κατοχώρες και στην Ιρλανδία. Θα πρέπει στα θεσμικά όργανα να διαμορφώσουμε την κοινή αποδοχή και ίσως να την υποστηρίξουμε και αυτό θα προσθέσει κάτι στις αποφάσεις που λαμβάνονται στο όνομα διαφόρων. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ρόλο να παίξει εδώ ως πλήρης Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, για να βοηθηθούν οι πολίτες. Ευχαριστώ. Τώρα έχει το λόγο η Επίτροπος Βάλστρομ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη. Ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση που νομίζω ότι θα μπορούσε να συνοψιστεί, αλλά για να γίνει αυτό θα επαναλάβω από τα όσα λέχθηκαν, ότι πρόκειται για ένα ουσιώδες στοιχείο της δημοκρατίας προτιμώ να το εξετάσω από την άποψη των πολιτών, τα δικαιώματα των πολιτών να γνωρίζουν τι συμβαίνει, να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, σε εγγραφά και να μπορούν ε, να παρακολουθούν και να μπορούν να επιλέξουν κατόπιν ενημέρωσης. Για όλους εμάς θα είναι ένα κρίσιμο έτος, διότι την 7η Ιουνίου οι πολίτες της Ευρώπης ε, θα ψηφίσουν. Και αυτό είναι ουσιώδες ε, νομίζω να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Έχουμε αναλάβει το βάρος ε, των διαφορών, ε, των διαφορών ανάμεσα στις κουλτούρες μας για το τι πρέπει να γίνεται γνωστό ή όχι. Εγώ έχουμε από μια χώρα που έχουμε μια μακρά ε, παράδοση της αρχής του ανοίγματο και της πρόσβασης στα έγγραφα, ενώ σε άλλα κράτη-μέλη είναι το αντίθετο. Έχουν μια παράδοση μυστικοπάθειας ε, και μόνο ότι δεν είναι μυστικό και απόρριτο καθίσταται δημόσιο, δημοσιοποιείται. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι έδειξε η εισήγηση της σχέσης της, ε, και της διασυνδέσεις ανάμεσα στα διάφορα αυτά θέματα και πρέπει να δούμε τα πράγματα από πολιτικής απόψεως. Η ομορφιά της συνθήκης της Λισαβόνας που θα διευρύνει αυτό το δικαίωμα ε, ενημέρωσης και πρόσβασης στα έγγραφα ε, και θα, θα κλείσει αυτό, θα δώσει ένα τέρμα σε αυτό το τυφλό παιχνίδι και ο κύριος Κάσμαν και άλλοι το ανέφεραν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ως στοιχείο για όλους μας. Νομίζω και ελπίζω ότι ε, μπορείτε να βασίζετε σε μένα για να αγωνιστώ σε καθημερινή βάση ούτως ώστε η Κομισιόν να βελτιώσει την πρόσβαση στα έγγραφα. Να δούμε τι γίνεται στις επιτροπές, στα μητρώα ορισμένα πράγματα που ανέφερε ο κύριος Καπάτο και μας βοηθούν. Θα πρέπει να κρατήσουμε την πίεση, να εξακολουθήσουμε να ασκούμε πίεση στην Επιτροπή, αλλά αυτό αναφέρεται επίσης και στο Κοινοβούλιο και μπορείτε να βελτιώσετε τα πράγματα και να συμβάλλετε στον άνοιγμα και στην διαφάνεια. Και αυτό είναι μέρος της ενίσχυσης της δημοκρατίας στην Ευρώπη και αυτό θα βοηθήσει στο να προετοιμαστούμε για τις ευρωεκλογές ε, που θα είναι και μια, μια σημαντική δοκιμή, δοκιμασία για όλους μας. Ευχαριστώ. Δίνω τον λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την ε, κυρία Επίτροπο. Ε, το είχα πει και προηγουμένως, αλλά η εισήγηση αναγνωρίζει ότι υπήρξε μια βελτίωση στην πρόσβαση στις ε, πληροφορίες. Υπάρχουν ε, πολλές απαντήσεις θετικές στα αιτήματα που λαμβάνουμε, αλλά πρέπει να αλλάξουμε και οπτική, διότι η πληροφορία πρέπει να υπάρξει για να δημοσιοποιηθεί δεν θα ήθελα να υπάρξει γραφειοκρατική επιβάρυνση σημαντική, υπερβολική. Αυτό που επιθυμώ είναι ένα σύστημα ε, το οποίο ήδη εξ ε, να υπάρχει, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση σε ένα έγγραφο όταν αυτό ζητείται, αλλά να υπάρχει και πρόσβαση στην πληροφορία όταν φτάνει αυτή, λαμβάνοντας βεβαίως τις υποχρεώσεις επιφύλαξης ως προς τις πολιτικές ομάδες και το λέω στο φίλο ε, Ντόιλ ε, διότι ο άλλος συνάδελφος έφυγε πρόκειται για μια διαθεσιμότητα πιο εύκολη των πληροφοριών πράγμα που δεν σημαίνει ότι δεν αφήνουμε στην ομάδα την ε, δυνατότητα να έχει συνεδριάσεις και κλεισμένων των θυρών. Δεν είναι μια πλήρης, μια απόλυτη υποχρέωση ολοκληρωτική. Πρόκειται για μια υποδομή που επιτρέπει τη διαφάνεια και νομίζω ότι αυτό που έλεγε ο συνάδελφος Σερό δεν είναι σωστό, δηλαδή ότι οι πληροφορίες για τις παρουσίες ε, και τις ε, ψηφοφορίες είναι όλες διαθέσιμες. Υπάρχουν τα πρακτικά ε, κάθε επιτροπής και οι πληροφορίες μπορούν να επιτευχθούν κάνοντας μια ερευνητική εργασία για κάθε συνεδρίαση. Εγώ ήμουν θύμα διότι μια ε, εφημερίδα ε, Ιταλική είπε ότι εγώ έχω τις περισσότερες απουσίες επειδή έφτασα στο, στα μισά της θητείας κάναν έναν υπολογισμό κατά τη διάρκεια ε, των μηνών που ήμουν παρόν σε σχέση με τα χρόνια που ήμουν απόν. Εμείς λοιπόν πρέπει να θέσουμε στη διάθεση του τύπου τις πληροφορίες για να επιτρέψουμε μια αναγνωσιμότητα σαφή, ούτω ώστε να αποφύγουμε τις χειραγωγήσεις και τις καταχρήσεις. Και ξέρω ότι η αξιοπρέπεια της κοινοβουλευτικής εργασίας δεν έγκυται στις απουσίες ή παρουσίες, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί εμείς πρέπει να κρύβουμε στο ίμιση αυτά τα στοιχεία, ανοίγοντας έτσι την πόρτα στις πιο δημαγωγικές καταχρήσεις και ελπίζω ότι για την άποψη αυτή όπως και για το θέμα ε, της πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες. Δεν ξέρω ε, γιατί το ΕΛΚΕ ζήτησε ξεχωριστή ε, ψηφοφορία γι' αυτό, αλλά ελπίζω ότι εδώ δεν θα έχουμε έκπληξη της τελευταίας στιγμής, διότι αυτό μου φαίνεται ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε για την ευελιξία σας. Ευχαριστώ κύριε Καπάτο, ελπίζω να επανεκλεγείτε. Έκλεισε η συζήτηση, θα έχουμε αύριο την ψηφοφορία. Συνεχίζουμε την ημερήσια διάταξη με την εισήγηση Λάμστορφ ε, για ε, το θέμα των προσφυγών για τα θέματα άμενας και ασφάλειας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν 13